Merci. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Push Up Brass Band των Βρυξελών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Good afternoon everybody. Thank you for coming. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρετίζει ο Πρόεδρος και στα γαλλικά. Σας καλωσορίζω στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Benvenuti a tutti Καλωσορίζω και όλους τους Ιταλούς, λέει ο Πρόεδρος στα Ιταλικά. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους δημάρχους από πόλεις που έχουν πληγεί από το σεισμό. Τους καλέσαμε ειδικά για να δείξουμε πόσο κοντά είναι η Ευρώπη στους πολίτες που αυτή τη στιγμή πλήττονται περισσότερο από άλλους. Συναποφασίσαμε με τους συναδέλφους του Προεδρείου, οι Αντιπρόεδροι και οι Κοσμήτορες να οργανώσουμε αυτή την μερίδα και να μετατρέψουμε την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα κοινοβούλιο των πολιτών. Σήμερα εσείς είσαστε εκείνοι που λαμβάνετε τις δικές μας θέσεις, που παίρνετε τη θέση μας. Είναι συμβολική αυτή η χειρονομία, αλλά ύψης της σημασίας γιατί δυστυχώς διανύουμε δύσκολους καιρούς με την τρομοκρατία. Είδαμε τι συνέβη τις προάλλες στο Ορλή, την παράνομη μετανάστευση, την οικονομική κρίση, η οποία πλήττει ιδιαίτερα πολλούς νέους που δεν μπορούν να βρουν εργασία. Αυτή τη δύσκολη στιγμή Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση προς τα θεσμικά όργανα, όπως είναι φυσικό, και έναντι της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Εμείς όμως θα θέλαμε το κοινοβούλιο αυτό στα επόμενα δυόμιση χρόνια και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που με συνόδευσαν σε αυτό το αξίδι. Θα θέλαμε λοιπόν να καλύψουμε αυτό το χάσμα μεταξύ θεσμικών οργάνων και Ευρωπαίων πολιτών. Θα θέλαμε εσείς που εκπροσωπείτε μισό εκατομμύριο πολιτών, 500 εκατομμύρια με συγχωρείτε πολιτών, να κατανοήσετε ότι εμείς προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Να σας εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε, ποιο είναι το έργο μας. Να μην είμαστε κλειστοί στα κτίρια των Βρυξελών, αλλά να είμαστε κοντά στους πολίτες, ανάμεσα στους πολίτες. Σήμερα γιορτάζουμε την 60η επέτειο της υπογραφής της ε, Συνθήκης της Ρώμης που έδωσε ζωή σε αυτή την Ευρώπη, που βεβαίως έχει πολλά ελαττώματα, όμως επέτρεψε σε πολλούς από μας, σε όλους, να ζήσουμε εν ειρήνη, με απόλυτη ελευθερία. Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα από μία πόλη στην άλλη, από μία χώρα στην άλλη. Είμαστε οι μόνοι, η Ευρώπη δηλαδή, όπου δεν ισχύει η θανατική ποινή. Σκεφτείτε τι γίνεται σε γειτονικέ χώρες που θέλουν να επανεισαγάγουν τη θανατική ποινή. Εμείς θέλουμε τα δικαιώματα του πολίτη και οι ελευθερίες του να είναι το κύριο μέλημά μας. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα, όχι μόνο για μία απλή διοργάνωση, αλλά για να κατανοήσετε ότι η Ευρώπη θέλει να αλλάξει, να γίνει καλύτερη αλλά χωρίς την Ευρώπη αυτή δεν θα φτάσουμε πουθενά. Πρέπει να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Δεν μπορούμε να καταστρέφουμε γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι σαν να αυτοτραυματιζόμαστε. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε τη στιγμή αυτή για να επιλύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα θα συζητήσετε και θα δείτε πώς εργαζόμαστε εμείς οι ευρωβουλευτές. Δεν είναι εύκολο να φτάσουμε σε σωστές ισορροπίες και λύσεις. Όμως σήμερα θα πειραματιστείτε άμεσα καθήμενοι στη θέση των ε, ευρωβουλευτών βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει και εκφράζοντας τις ιδέες σας κανένας δεν, θα σας απαγορεύσει να μιλήσετε. Ενώ σε άλλες ε, πλευρές του κόσμου συμβαίνουν πολλά δεινά, μπορείτε εσείς να επικρίνετε την Ευρώπη ή τους ευρωβουλευτές, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά το λέτε ελεύθερα. Μιλάμε για αξίες, για τήρηση των αξιών. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η Ευρώπη. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Η πρώτη αντιπρόεδρος θα αναλάβει την συνεδρίαση αυτή, η κυρία Μακίνες, που έχει μεγάλη πείρα, προέρχεται από την Ιρλανδία. Θα δείτε ότι όλοι μιλάμε διαφορετικές ε, γλώσσες, αλλά έχουμε την ίδια ταυτότητα. Ακούσατε και την Πούσα Brass Band, η οποία εξέφρασε την Ευρώπη με μουσική. Πρόκειται για μία κοινότητα ιδεών και αξιών. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν και την πανηγυρική συνεδρίαση της Ρώμης που πιστεύω ότι θα είναι μια στιγμή μιας νέας όθησης και πνοής για την Ευρώπη, πιστεύω ότι γυρνώντας στην πατρίδα σας θα μπορέσετε να αφηγηθείτε αυτή την ημέρα το τι αισθανθήκατε, το ότι σε μια μεγάλη δημοκρατία μπορεί κανείς να μιλήσει ελεύθερα και υπάρχουν 751 ευρωβουλευτές που σας θεωρούν πρωταγωνιστές και που πρέπει να εργαστούν για σας και να σας δώσουν απαντήσεις. Πριν δώσω το λόγο στην πρώτη αντιπρόεδρο, στην κυρία Μαγκίνες, θα ήθελα το κορίτσι που κάθεται δίπλα μου να καθίσει στη θέση μου για να δείτε πώς και ένας νέος, μία νέα μπορεί να προεδρεύσει. Για να δείτε, για να δείτε πόσο υπεύθυνοι είναι και οι νέοι. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Έλα να καθίσει στη θέση μου. Η Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας ε, καλωσορίσατε εδώ, που υποστηρίζετε την ε, νεότητα, την νεολαία και τους εκπροσώπους και δίνω το λόγο στην κυρία Μαγκίνες. Um, θα ήθελα απλά να πω κι εγώ ότι πολύ ευχαρίστω ε, να συνεχίσετε να προεδρεύετε στη συνεδρίαση, αν το θέλετε βέβαια. Ε, εν περιπτώσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταγιάννη για τις, τα θερμά του λόγια, τα λόγια με τα οποία σας καλωσόρισε, πολύ ζεστά και θερμά λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε επίσης που σκεφτήκατε ακριβώς αυτό, το να φέρετε τους πολίτες στα δικά μας τα έδρανα. Ελπίζω λοιπόν να το ευχαριστηθείτε και να συμμετάσχετε στις σημερινές διαδικασίες. Εγώ έχω ένα πολύ δύσκολο καθήκον. Ξέρετε, το να τηρούμε το χρόνο, αυτό που κάνουμε και στην Ολομέλεια και θα είμαι πολύ αυστηρή. Έχουμε πέντε θέματα να εξτάσουμε πολύ σοβαρά. Η νεολαία και η παγκοσμιοποίηση, η Ευρώπη των 27 και το μέλλον, η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και το πλαίσιο είναι το εξή ότι ε, θα έχουμε μία εισήγηση ως εναρκτήριο ομιλία ε, από τα μέλη βέβαια του Κοινοβουλίου που είναι σήμερα κοντά μας και μετά μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις και ε, να έχετε βέβαια και τον αριθμό σας για να μπορούμε να τον βλέπουμε και εμείς. Ο λόγος γιατί είναι μεγάλη αυτή η αριθμή είναι γιατί εγώ δεν βλέπω καλά. Φοράω βέβαια γυαλιά, αλλά δεν βλέπω και τόσο καλά. Ελπίζω να σας δω όταν θα σηκώσετε τον αριθμό σας ε, και σας παρακαλώ να μην ζητήσετε όλοι μαζί το λόγο. Δεν γίνεται αυτό, αλλά χαίρομαι που έχετε τους αριθμούς και αυτό σίγουρα θα διευκολύνει ε, το να σας ε, βλέπω. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πολλοί θέλουν να λάβουν το λόγο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο θέμα είναι η ανεργία των νέων και η πρόκληση για την Ευρώπη το να προσφέρει εργασιακές ε, ε, ευκαιρίες σε όλους. εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο επ' αυτού. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Τίνα Χόκοβα, μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ε, σήμερα ε, κατ' ουσίαν εκπροσωπώ εκατομμύρια νέους από ολόκληρη την Ευρώπη και σας στέλνουμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι ε, περισσότεροι νέοι να βρουν θέση απασχόλησης και εδώ πρέπει να εφαρμόσουμε δύο λύσεις. Πρώτον, να μην υπάρχουν αποκλεισμοί, η απασχόληση ε, να μην έχει κανένα αποκλεισμό, να στηρίζει όλους τους νέους και κυρίως να απευθύνεται στις πιο ευάλωτες ομάδες. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τρεις συμπληρωματικές πράξεις. Πρώτον, ένα ε, πρόγραμμα για τους νέους, εγγύηση για τους νέους, χωρίς αποκλεισμούς, προσαρμοζεται στους νέους, με συγκεκριμένες ανάγκες, νέες γυναίκες, νέα ε, αγόρια. Αυτό να είναι προσπελάσιμο για όλους τους νέους. Μετά, μόνο απευθυντικές θηρίδες, τα one-stop shop όπως είναι γνωστά, να έχουν όλοι καθοδήγηση στον ίδιο χώρο και έτσι να στηρίζεται η μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Και τέλος, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να παραλείψουμε τη δράση. Τη δράση με τους βασικούς μας εταίρους να συμμετέχουν οι οργανώσεις νεολαίας. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για να έχουμε πρόσβαση στους πλέον ευάλωτους νέους. Γιατί οι οργανώσεις νεολαίας έχουν μεγάλη διαδικτύωση, δουλεύουν είναι στη βάση, είναι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν την καθημερινότητα. Αυτοί λοιπόν μπορούν να γύρουν γέφυρες με τους νέους και με τις υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Δεύτερη λύση, δίκες συνθήκες απασχόλησης ανεξάρτητα από τη μορφή της απασχόλησης. Πώς μπορούμε άραγε να το πετύχουμε αυτό με ε, κοινωνικά δικαιώματα τα οποία θα είναι εγγεγραμμένα σε όλα τα συμβόλαια απασχόλησης και στα επισφαλή να δουλέψουμε με την πλατφόρμα της οικονομίας και με άλλες μορφές απασχόλησης. Ελάχιστες εγγυήσεις για τους εργαζόμενους συμπεριλαμβανομένου και του σωστού μισθού όπως και η δυνατότητα να συμμετέχει κανείς σε συνταξιωτικά προγράμματα. Και τέλος, ίση αμοιβή για ίδια εργασία. Δεν μιλάω εδώ για τις διαφορές ανάμεσα στα φύλλα, αλλά εγώ εκείνο που λέω είναι ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν διακρίσεις με βάση και την ηλικία. Ε, εμείς λοιπόν ε, από το φόρουμ της νεολαίας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με εσά. Ελπίζω μαζί να διανύσουμε τον δρόμο που οδηγεί στο μέλλον και ξεκινάμε τώρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το εναρκτήριο λάκτισμα στην ομιλία. Καλό λοιπόν την κυρία Στάνρουκ από τους σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ να λάβετε το λόγο και να απαντήσετε σε δύο λεπτά. Θα είμαι πάρα πολύ ε, απλή, απλά ε, υπογραμμίζω, συμφωνώ και παυξάνω με όλα αυτά που είπε η Τίνα. Και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι σοσιαλδημοκράτε, αγωνιζόμαστε υπό την καθοδήγηση του κυρίου Πιτέλα. Αγωνιζόμαστε για καλέ θέσει απασχόληση, για την αντιμετώπιση τη ανεργία, κυρίω τη ανεργία των νέων. Το 2012 έχουμε την εγγύηση, το μέσο εγγύηση για του νέου. Το φέραμε αυτό στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτό το μοντέλο επιτυχία ήδη καρποφορεί. Πάρα πολλοί νέοι με αυτό το εργαλείο έχουν βρει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εξάλλου αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και οι συνθήκες εργασίας. Οι νέοι πρέπει να αμείβονται όταν εισέρχονται στην αγορά εργασία, όχι απλήρωτες θέσει δοκιμαστική εργασία για τους μαθητευόμενους. Επίση, τα one-stop shop είναι πολύ σημαντικά ε, να υπάρχουν καλά πρότυπα, Έχουμε πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη. Εξάλλου η Ευρώπη έχει την ευκαιρία όλα αυτά τα καλά παραδείγματα από διαφορετικές χώρες αυτά να τα μεταφέρει σε άλλες χώρες όπου επίσης υπάρχουν προβλήματα για να δείξει πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί παραδείγματος χάνει το πρόβλημα μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Κάθε νέος ο οποίος έχει χάσει κάποια στιγμή την ευκαιρία να μπει στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζει προβλήματα διαβίου. Αυτό το βλέπουμε από στοιχεία που αφορούν στο παρελθόν και οι αρχέ του να βρίσκει κανεί θέση απασχόληση στον ίδιο χώρο που ζει. Αυτό θα έλυνε πολλά σημαντικά προβλήματα, θα προήγαγε την κοινωνική σύγκληση. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω αυτά που είπε η Τίνα. Βεβαίω και τη στηρίζουμε, βεβαίω και στηρίζουμε όλου του νέου τη Ευρώπη. Για μα ε, οι νέοι είναι προτεραιότητα τη πολιτική μα. Πριν δώσω το λόγο ε, στον επόμενο συνάδελφο, να μην ξεχνάτε ότι θα δεχτούμε ερωτήσει. Όποιο θέλει να υποβάλει ερώτηση, να σηκώνει τον αριθμό του. Κάθε φορά θα έχουμε τέσσερι ερωτώντε. Και τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να σηκώσετε τον αριθμό, να δείξετε ότι θέλετε να υποβάλλετε ερώτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λοπέζε, η οποία είναι από την Ενωμένη Αριστερά. Παρακαλώ, δύο λεπτά παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω, εσάς τους νέους, τους πολίτες της Ευρώπης. Εδώ είναι το σπίτι σας. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Σημερίζομαι την άποψη της ε, εισηγήτριας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την σωστή και δίκαιη εργασία για τους νέους. Και συμμερίζομαι αυτά που προϋπόθηκαν, δηλαδή από πλευράς Ευρωπαϊκής Αριστεράς θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεισφέρουμε όχι μόνο με προγράμματα εγγύησης για τους νέους, αλλά και με άλλες πολιτικές που να σχετίζονται με τις αλλαγές στα πρότυπα παραγωγής τα οποία ισχύουν σήμερα. Θεωρούμε ότι η πολιτική λιτότητας δεν μπόρεσε να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε και έχουμε προβάλει εναλλακτικές λύσεις για να επιληθούν τα θέματα των νέων συνεργαζόμαστε για τον κοινωνικό ευρωπαϊκό πυλώνα, αλλά και για την κατάρτιση και εγκρίναμε πρόσφατα το EURES που είναι ένας μηχανισμός κινητικότητας για τους νέους καθώς και το συντονισμό των δημοσίων αρχών για την εργασία. Δυστυχώς στην Ευρώπη υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να βρούμε ένα εργασιακό πλαίσιο για να μπορέσουμε να κινηθούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Τώρα θα έρθουμε στους ομιλητές μας. Το πρώτο πρόσωπο είναι το 247. δείτε τον αριθμό του. Δηλαδή, είναι ο αριθμό 247. Παρακαλώ να σηκωθείτε πράγματι. Πρόκειται για μια ευτυχή σύμπτωση. Δεν έγινε επίτηδε. Τη γνωρίζω την κυρία και είναι Ιρλανδή όπω. εγώ. Πολύ ευχαρίστω να σας δώσω πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leader που ε, κλείνει 25 χρόνια τώρα. Και ήταν πιθανώς το πρώτο πρόγραμμα το οποίο έφερε την Ευρώπη σε άμεση επαφή με τους πολίτες της που ζουν στην Ήπεθρο. Θέλω να ζητήσω αυτό το πράγμα που είναι το αποκορύφωμα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας που στηρίζει και διασφαλίζει να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό, να φροντίσετε να συνεχίσει να μείνει στα χέρια των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των τοπικών κοινοτήτων. Να παραμείνει δηλαδή ένα δυναμικό πρόγραμμα το οποίο θα αφαιρεί τους νέους αλλά και τους ηλικιωμένους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσουν τα μέλη μας, οι ευρωβουλευτές δηλαδή, πολύ σύντομα μετά. 197. Είναι ο επόμενο αριθμό που έχει λόγο. Είμαι ο Μπερνάρντο Ράμος από την Ισπανία. Συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Ομοσπονδιακό Σχήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνετε. Εγώ είμαι πατέρας δύο νέων παιδιών με πανεπιστημιακές σπουδές οι οποίοι είναι άνεργοι και χωρίς καμία ελπίδα εξέβρεσης εργασίας. Στην ατζέντα σας υπάρχει και το θέμα της ανεργίας των νέων. Αλλά είμαι κάπως απογοητευμένος γιατί βλέπω ότι το αντιμετωπίζετε από πλευράς συμπτωμάτων και όχι αιτιών. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βοηθήσει αυτή την ευρωπαϊκή κοινωνία και να κατέχει και ηγετική θέση. Σήμερα δεν δημιουργείται πλούτος ανά τον κόσμο, ενώ υπάρχει μεγάλη δυνατότητα προς αυτή την κατεύθυνση εξαιτίας των τεχνολογιών εχμής. Χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Βρισκόμαστε ενώπιον συνταρακτικών αλλαγών, είτε το θέλουμε είτε όχι. Μπορεί να είναι τραυματικές αυτές οι αλλαγές, αλλά θα ήθελα εσείς ως πρωτοπόροι να προτείνετε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση και να μην πρέπει να την υποστούμε στο δίνεκες. Now, ευχαριστώ πολύ. 548. 548 είναι ο επόμενος αριθμός. 548. I can't see. You got to stand. Ah. Α, τώρα σας είδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, σας βλέπω. Σας βλέπω. Ε, βεβαίως. Ευτυχώς είδα και το νούμερο. Πρέπει να βλέπω και προς την κατεύθυνσή σας. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα, είμαι ο Σέρτζο Καραμάτσα και έρχομαι από την Φαβάρα, μια περιοχή στο Αγριτζέντο, στην τόσο όμορφη Σικελία. Σήμερα αναφέρεται στην μέση διάταξη η ανεργία των νέων. Ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο να υπάρχει με τον ίδιο τρόπο και την ίδια μορφή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το ξέρουμε κυρίω εμεί, οι νέοι του νόου. Αυτό όμω που απασχολεί είναι κάτι άλλο. Θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σα σε ένα στοιχείο τη ανεργία των νέων που ποτέ δεν το έχετε εξετάσει. Αναφέρομαι στην ανεργία στην επαρχία, στην επαρχία της Ευρώπης, ε, στην Ήπετρο της Ιταλίας, ε, στις ε, περιοχές που είναι μακριά από το κέντρο. Σε αυτές τις περιοχές η ανεργία των νέων είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα από ό,τι στις μεγάλες πόλεις. Και εκπροσωπώ νέους που έρχονται από πολλές περιοχές, από την Ήπετρο Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, τι είδους Ευρώπη επιθυμούμε, τι θέλουμε να γίνει με την Ήπετρο, Εγώ πιστεύω ότι η Ήπετρος είναι πεμπτουσία σημασία των ευρωπαϊκών κρατών και δεν πρέπει να πετάνε. Για να μείνουν εκεί οι νέοι ε, θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, να τους εγγυηθούμε την εργασία που θα συνδέεται με τη γη και που θα τους διασφαλίζει και τη ζωή στην ίδια τη γη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο... 300... Αριθμός 350. 350. Καλό σας απόγευμα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας καλέσατε εδώ. Ονομάζομαι ε, Λορένα Ράμος και εργαζόμαστε για να υπάρχουν, να προωθηθούν προγράμματα πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Θέλουμε να προωθήσουμε την απασχόληση εγκάρσια σε όλους τους τομείς, τους τομείς όπου να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μεγάλο μισθολογικό χάσμα, το οποίο μειώθηκε όμως μεταξύ 2007 και 2015. Όμως υπάρχει υψηλή ανεργία και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερη ανεργία έναντι των ανδρών. Εργαζόμαστε σε προσωρινές εργασίες με χειρότερες συνθήκες και χειρότερη πληρωμή. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε παρά να απευθυνθούμε στον Πολωνό Ευρωβουλευτή, ο οποίος ε, μίλησε κατά απαράδεκτο τρόπο κατά των ε, γυναικών. Δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι γυναίκες ε, είναι και αυτές που συνεισφέρουν και αποτελούν πηγαίο ταλέντο της κοινωνίας. Thank you. Η κυρία Μακίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα αυτά, αυτά λοιπόν είχαν ε, σχέση με ισότητα, ανάπτυξη της υπαίθρου, των κοινοτήτων της Υπέθρου, καθώς και την ανάγκη για ένα νέο οικονομικό πρότυπο. Μπορείτε εσείς, κυρία Στάνιερ, να μιλήσετε για ορισμένα από αυτά τα θέματα. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά είναι πολύ λίγος χρόνος. Πράγματι όλα τα προγράμματα τα οποία απευθύνονται στους πολίτες και τις πολίτες της Ευρώπης είναι, ισχύουν για όλους, σε όποιο τομέα της πολιτικής και αν αναφέρονται. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα προγράμματα αυτά, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα Leader. Πράγματι, ο πατέρας των δυο νέων που έχουν ολοκληρώσει τις ε, πανεπιστημιακές τους σπουδές, τα παιδιά του δεν είναι δυστυχώ μεμονωμένη περίπτωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Υπάρχει και το πρόγραμμα εγγύηση για την νεολαία άνθρωποι που βρίσκονται χωρίς απασχόληση μετά από τις σπουδέ τους, θα έχουμε υπόψη μας αυτά τα πράγματα. Όμως η ανεργία μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο επί τόπου, με επενδύσεις. Επί τόπου, ξαναλέω. Και αυτό ισχύει και για τις περιοχές της Υπέθρου. Μόνο έτσι μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Όπου έχουμε σημαντική ανεργία, έχουμε και σημαντική ανεργία των νέων. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Καμία περιφέρεια να μην αιμορραγεί στην Ευρώπη, να μην φυκώνονται να φεύγουν οι νέοι για να πάνε εκεί όπου υπάρχουν θέσεις εργασίας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να μπει ένα τέρμα στην πολιτική λιτότητα, να ενισχυθούν οι επενδύσεις, να ενισχυθεί η οικονομία επιτόπου για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ανεξαρτήτως του αν ο νέος ή η νέα έχει το απολυτήριο του σχολείου ή το πτυχίο του πανεπιστημίου. Επίσης για μας η ενίσχυση της θέσης των γυναικών αλλά και το άνοιγμα δυνατοτήτων στην απασχόληση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί όχι μόνο για την ανεργία, αλλά και για την ισότητα των γυναικών. Πολλές γυναίκες ζουν σε εντελώς αβέβαιες, εντελώς επισφαλείς συνθήκες, γιατί έχουν και επισφαλείς θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί και όχι μόνο για την επέτειο ε, των δικαιωμάτων των γυναικών. Για όλους μας απασχολεί αυτό. Θα συνεχίσουμε από την Ευρώπη να δίνουμε κίνητρα για την θέσπιση ισότητας γυναικών και ανδρών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρώπη φρόντισε να γίνουν τα πράγματα αυτά πραγματικότητα και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για αυτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Λόπεζ, δύο λεπτά παρακαλώ. <laughs> Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις και να κάνω ορισμένα σχόλια. Έγινε λόγος για τα προγράμματα αυτά, τα οποία θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, όπως το μέσο για τους νέους ή ο ορίζοντας 2020 μεταξύ άλλων. Αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη κατανομή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και ιδιαίτερα ποιοτική εργασία για τους νέους. Ο κύριος Μπερνάρδο είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σωστό. Θα πρέπει να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές, όπως είπατε. Χρειάζεται μία μετατόπιση των πολιτικών μας, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από μία κατάσταση κλειδονισμών και κρίσης που ζούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ξεχωριστές πολιτικές, μία οικονομική και μία κοινωνική, είναι αλληλένδετες. Ως προς τα ε, θέματα ισότητας των δύο φύλων και την Ήπεθρο, καταρχήν στην Ήπεθρο θα πρέπει να παραμένουν οι κάτοικοι εκεί με κίνητρα και να υπάρχουν οι ίδιες υπηρεσίες στην Ήπεθρο με τα μεγάλα αστικά κέντρα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, ιδιαίτερα στο νότο της Ευρώπης. Βεβαίως, στις αγροτικές περιοχές μπορεί κανείς να ζει με έναν αξιοπρεπή μισθό γιατί τα προϊόντα πολλούνται στη σωστή του τιμή χωρίς μεσάζοντες και έτσι οι νέοι και οι νέοι αγρότες μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους. Έχουμε μεγάλο έλλειμμα γυναικών και νέων στις αγροτικές περιοχές και γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Γνωρίζω ότι αυτό το θέμα το χειριζόμαστε επιφανειακά κάπως λόγω έλλειψης χρόνου. Πόσοι θεωρείτε ότι η, ότι η Ευρώπη κάνει κάτι για τους νέους και για την ανεργία των νέων. Πόσοι πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει το θέμα της ανεργίας των νέων. Ναι, δείχνετε το επίπεδο της απογοήτευσής σας και ελπίζω κάποιος να πάρει μια φωτογραφία της απάντησης σε αυτό το ερώτημα γιατί είναι ενδεικτική. Επόμενο θέμα, το οποίο δημιουργεί διχασμούς ως προς την παγκοσμιοποίηση και το σωστό επιμερισμό καθηκόντων. Πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι πολύ οι ευεργετημένοι από την παγκοσμιοποίηση. Η Νατάλια Αλόνσο έχει το λόγο από την Oxfam. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία σκέψη για να το σκεφτείτε λιγάκι. Γνωρίζετε πόσοι άνθρωποι κινδυνεύουν από φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το σκεφτείτε λιγάκι και πιστεύετε ότι η Ευρώπη είναι από τις πιο πλούσιες υπήρους, ε, τι θα λέγατε, ένα στους δέκα, δύο στους δέκα. Η αλήθεια, η πραγματικότητα είναι ότι ένας ε, κάθε τέταρτος, κάθε τέταρτος πολίτης, 103 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κινδυνεύουν από τη φτώχεια και παράλληλα η Ευρώπη φιλοξενεί 342 δισεκατομμυρίχους. Η φτώχεια και η ανισότητα δεν είναι κάτι το σπάνιο και είναι και πολιτική επιλογή. Πρώην πρόεδρος Ομπάμα είπε ε, ένα κόσμο, σε ένα κόσμο όπου το 1% κυριαρχεί πάνω στο 99%, είναι ένα ασταθής κόσμος. Η παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να ισχύει για όλους και όχι μόνο για λίγου. Όταν έχουμε έναν κόσμο όπου Πολύ λίγοι κατέχουν ε, πολύ περισσότερα από όλου του φτωχού. Κάτι δεν πάει καλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα παγκόσμιο ε, παίκτη και έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στο να στηρίξει τι αναπτυσσόμενε χώρε για να εξαλείψουν η φτώχεια, αλλά επίση και για να διασφαλίσει ότι όλε οι ενωσιακέ πολιτικέ συμβάλλουν προ αυτή την κατεύθυνση. Πώ μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα. Πρώτα απ' όλα με τι φορολογικέ πολιτικέ. Πρέπει να ανακατανεμηθεί ο πλούτο, να μειωθεί η φτώχεια επίσης οι εταιρείε να συμμετέχουν σε αυτό που τους αναλογεί και οι κυβερνήσεις να έχουν τα χρήματα για να προσφέρουν υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίσει ότι οι εταιρείε θα λογοδοτούν πώς προσπορίζονται τα κέρδη και πώς ακριβώς κατανέμουν τα κέρδη αυτά. Ένα άλλο πράγμα στο οποίο μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λειτουργήσει σωστά η παγκοσμιοποίηση είναι η μετανάστευση. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφέ ότι η μετανάστευση μπορεί να είναι επωφελή ε, και, ε, και για αυτού που μεταναστεύουν και για τι φιλοξενούσε χώρε. Οι μετανάστε έχουν στείλει διπλάσια ποσά στι αναπτυσσόμενε χώρε από τα χρήματα που έλαβαν οι χώρε μετανάστευση. Άρα δηλαδή νέο αφήγημα, ένα αφήγημα που θα προβλέπει ευκαιρίε και γι' αυτό η Oxfam θέλει να υπάρχει η ανθρώπινη οικονομία όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο των αποφάσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Κασπάρη από το ΕΛΚΑ για να απαντήσει. Παρακαλώ, Ντάνιελ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί πολίτες, η παγκοσμιοποίηση υπάρχει και βρισκόμαστε μπροστά στην ε, δυνατότητα είτε να συμμετέχουμε είτε να απέχουμε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία χώρα που δεν συμμετέχει στην παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι η Βόρεια Κορέα. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκεί ε, έχουν μία τραγική μοίρα, αυτό οφείλεται στο ότι βιώνουν έναν ε, στιγερό δικτάτορα, αλλά και στο ότι είναι απομονωμένοι. Εάν λοιπόν θέλουμε να συμμετέχουμε, πρέπει να συνδιαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση. Και ζούμε σε ένα κόσμο όπου ε, στις ε, πατρίδες μας αποφασίζουν σε τοπικό επίπεδο οι δήμοι και οι κοινότητες, κατόπιν σε εθνικό επίπεδο τα κοινοβούλια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Όμως ένας, ε, μια κυβέρνηση που να θεσπίζει κανόνες για ολόκληρο τον κόσμο δεν υπάρχει. Άρα δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα η παγκοσμιοποίηση είτε να καθορίζεται από τους πιο πλούσιους, τους πιο άδικους, τους πιο γρήγορους, τους πιο πονηρούς ή έχουμε την ευκαιρία εμείς να συνδιαμορφώνουμε την παγκοσμιοποίηση όπου ως διεθνής κοινότητα καθορίζουμε κανόνες και αυτό είναι εκείνο το οποίο εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια είτε με τις εταιρικέ μας συμφωνίες είτε με τις συμφωνίες μας για το εξωτερικό εμπόριο. Έχουμε ρυθμίσει πάρα πολλά θέματα ε, ας πούμε για το πώς λειτουργούν οι οικονομικές σχέσεις και πριν από λίγες μόνο εβδομάδες εμείς καθορίσαμε και επιβεβαιώσαμε τις εμπορικές μας σχέσεις με τον Καναδά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομιλώ βέβαια μόνο εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς με το 1 τρίτο των Ευρωβουλευτών είμαστε η πιο ισχυρή πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλουμε διεθνείς συμφωνίες, εφαρμόσιμες. Εγώ όμως δεν θέλω να αναφέρουμε μόνο τους αρνητικούς αριθμούς όπως ακούσαμε για τη φτώχεια. Η παγκοσμιοποίηση κατόρθωσε στην Ασία, στην Κίνα, ε, εκατομμύρια ανθρώπους να τους απελευθερώσει από τη φτώχεια. Και στην Ευρώπη πολύ πολίτες εποφελούνται από χαμηλές τιμές και καλέ θέσει απασχόλησης. Άρα δηλαδή συνδιαμορφώνουμε την κοσμιοποίηση. Εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματα και τότε βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο στην κυρία εκ δεξιών σας, ε, στην κυρία Σάκα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Oh. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι εξαιρετική ευκαιρία να καλωσορίζω όλους εσάς εδώ. Ε, χαίρομαι που εσείς φέρατε και τη μουσική μαζί σας, γιατί δεν την έχουμε πάντα εδώ. Είναι καλό να πανηγυρίζουμε για αυτά που έχουμε επιτύχει. Βεβαίως ξέρουμε για τη φτώχεια και τις ανισότητες ανά τον κόσμο. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά Μερικές φορές ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην Ευρώπη έχουμε πολύ υψηλή ποιότητα ζωής και να την κρατήσουμε. Οι συνάδελφοι το προανέφεραν, υπάρχει ανάπτυξη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομική ανάπτυξη δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήνουμε τους άλλους ε, στην άκρη, αλλά είναι και κάτι το θετικό. Δεν θέλουμε να κάνουμε έναν αγώνα προς τα κάτω μέσα στα πλαίσια της ε, παγκοσμιοποίησης, γιατί πολλές φορές οι μεγάλες πολυεθνικές επιδιώκουν και τα μεγαλύτερα κέρδη. Θέλουμε σαφείς κανόνες που να μας διέπουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε την οικονομία μας. Δηλαδή, αν θέλουν να εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να τηρούν ορισμένες προδιαγραφές. Να προστατεύσουμε επίσης και το περιβάλλον, την ασφάλεια των καταναλωτών και φυσικά έτσι να επηρεάσουμε με όλο το οικονομικό μας βάρος. Είναι πάντα εφικτό όχι πάντα. Γίνονται όμως πολλές συζητήσεις για το ποιο χαρακτήρα πρέπει να έχει το εμπόριο και χαίρομαι διότι αυτή η, ζω... η ζωηρή συζήτηση οδήγησε σε μια νέα ατζέντα, σε μια νέα εμπορική πολιτική μέσα στα πλαίσια των ε, αξιών της Ευρώπης. Ονομάζεται Trade for All το οποίο σημαίνει ότι δεν θέλουμε να πολεμήσουμε την παγκοσμιοποίηση, γιατί δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, αλλά θα πρέπει να διέπεται από κανόνες η παγκοσμιοποίηση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες με λιγότερη ανισότητα. Έχουμε δύο μιλητές. 424. Έχετε το λόγο. parlement. Goedemiddag ehm, Καλό σας απόγευμα. Απευθύνομαι σε όλους τους παρόντες και βεβαίως και τους ευρωβουλευτές. Λέγομαι Ντεβίλες και είμαι Βέλγος από την Αμβέρσα. Με το τρένο μία ώρα προς βορρά από τις Βρυξέλλες. Με συγχωρείτε μια ωρα προς απο Είναι καλύτερο να κρατάτε κάποιο, κάποια μικρή απόσταση από το μικρόφωνο, ας πούμε ε, περίπου ε, μισό μέτρο. Ακούγεται πολύ καλύτερα τότε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, καλό σας απόγευμα αγαπητές και αγαπητοί ευρωβουλευτές, εσείς κυρία Πρόεδρε, λέγομαι Ντεβίλερς και έρχομαι από την Αμβέρσα που είναι μια πόλη βελγική, μια ώρα περίπου με το τρένο από εδώ, από την Ένωση Ευρωπαίων Σπουδαστών της Αμβέρσας και είμαστε μέλος της ε, Ένωσης Stand Up for Europe. να, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζετε ότι οι πλουσιότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη πληρώνουν μόνο 2% φόρους. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε ώστε οι επιχειρήσεις να καταβάλουν τους φόρους τους εκεί όπου παράγεται και πωλείται το προϊόν τους. Αυτό πρέπει να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς διατρέχουμε όλοι τον κίνδυνο οι χώρες να στραφούν οι μεν κατά τον δε και αυτό να εξυπηρετεί μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το βάλουν ως στόχο οι Students for Europe και θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση από εσά. Βλέπω πολύ έντονη υποστήριξη για την ερώτησή σας. Ε, θα ήθελα να δω αριθμούς 426 και μετά 104. 426. 426. Καλό σας απόγευμα και από μένα. Λέγομαι Μπράνι και εγώ μιλώ εξ ονόματος των Students for Europe της Αμβέρσας. Νομίζω η παρατήρηση του συναδέλφου μου μόλις μίλησε ήταν ορθή και δικαιολογημένη. Έχει προκληθεί ένα κλίμα φόβου. Οι άνθρωποι δεν έχουν πια το θάρρος να προχωρήσουν στην ίδρυση επιχειρήσεων. Έχει εκλείψει το επιχειρήν. Πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε οι άνθρωποι να παρακινηθούν να επιζητήσουν και πάλι τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Ορίστε εσείς παρακαλώ 104. Λέγομαι Ζαν Λουί Ρωσινιό, απλός Ευρωπαίος πολίτης. Συνεχίζω από τις ερωτήσεις που έκαναν οι δύο νεαροί προηγουμένως. Έχω μια συνολικότερη ερώτηση. Υπάρχει μια εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι ικανή να λέει μόνο «Κοιτάξτε, θα έπρεπε να κάνετε αυτό ή θα έπρεπε να κάνετε εκείνο». Χωρίς όμως ε, να έχει καμία περιοριστική δυνατότητα και αποφασιστική αρμοδιότητα ε, στα μέλη της. Η ερώτησή μου λοιπόν και νομίζω η ερώτηση αυτή τίθεται πραγματικά στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό ανάμεσα σε αυτά που ακούμε και σε αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη γνώμη σας γι' αυτό. Η σας ευχαριστώ πολύ. Εκατόν σαράντα. σαράντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ είμαι δήμαρχος από την Τέρα στο Αμπρούτσο και από κοινού με τους άλλους δύο συναδέλφους εκπροσωπώ την κεντρική Ιταλία. Την Ιταλία εκείνη που μαρτύρησε από το σεισμό, από τις χιονοθύελες, από τις κατολιστήσεις. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την εργασία, για την ασφάλεια, για την απερίμωση των, ε, της υπαίθρου και αυτό που βιώνουμε είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες, διότι οι δικοί μας οι πολίτες εγκαταλείπουν τις πόλεις μας, ε, τα παιδιά μας, ε, αν δεν γίνει κάτι, δεν τα έχουν μέλλον. Εμείς λοιπόν ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε τη βοήθεια της Ευρώπης, ε, που κάνει βέβαια πολλά για μας, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερα, να είναι ακόμα πιο κοντά μας, γιατί αυτό που έγινε στη δική μας περιοχή ήταν κάτι το απρόβλεπτο, μια έκτακτη κατάσταση, άρα είναι απαραίτητο να υπάρχουν υπάρχουν και έκτακτα μέτρα. Το ζητήσαμε από την κυβέρνησή μας, από την περιοχή μας, τώρα το ζητάμε και από την Ευρώπη μας. Γιατί η Ευρώπη έχει και καλή κατοίκους στο Αμπρούτσο, στο Λάτσιο, Θέλουμε λοιπόν ε, να αποδείξει η Ευρώπη ότι είναι η μαμά αυτών των περιοχών. Και είμαστε εδώ για να το ζητήσουμε αυτό και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ταγιάννη που μας έδωσε δυνατότητα να έρθουμε. Εμείς είμαστε δήμαρχοι που κάθε μέρα έρχονται αντιμέτωποι με τις ε, δυσκολίες του να ζουν οι άνθρωποι σε περιοχές ε, σεισμόπληκτες με λίγα σχολεία. Ε, έχουμε μια περιοχή σε κρίση, μαγαζιά που κλείνουν, οικονομία που έχει γονατίσει. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για την περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και πραγματικά ε, νιώθουμε μεγάλη ε, συμπάθεια και έντονα συναισθήματα με εσά και την περιοχή σας. Λοιπόν, ε, θα σπάσω τον κανόνα, θα πάρουμε και μια πέμπτη ερώτηση. Και μου επιτρέπετε να το κάνω αυτό. Το 159 παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη, ο κύριος με το 159. Ah, euh, bonjour à tous. Euh, Δεν θα ήθελα να ε, υποβάλω μία ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κάσπερη για την παγκοσμιοποίηση. Ξέρουμε ότι δημιουργεί μεγάλα ερωτήματα ως προς την οικονομία, ως προς την κοινωνία, πολιτισμικά και ούτω καθεξής. Και βλέπετε αυτά τα τεράστια ερωτήματα που απασχολούν όλους μας εδώ στην Αφρική, στο Μπαγκόκ, σε όλες τις πλευρές και σημεία της γης. Εάν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση ε, κατάματα, δεν θα τα καταφέρουμε. Μιλήσατε για την Βόρειο Κορέα. Δηλαδή είπατε ότι η μόνη εξαίρεση είναι η Βόρεια Κορέα. Αυτό το θεωρώ αθέμητο και εδώ είναι το ζήτημα που θέτω. Είναι σαν να θέλετε να μετατοπίσετε την ουσία του ζητήματος. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης. Εγώ ε, μπορώ να σας πω πότε πρωτοείδα την Ευρωπαϊκή Σημαία. Είναι κάτι που με συγκίνησε. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι συμβολισμοί να είναι εύστοχοι και να αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Είδαμε στη Γαλλία τι έγινε με τα αποτελέσματα των εκλογών και δεν αφορά ε, μόνο την άκρα δεξιά. Φαίνεται ότι πολλοί νέοι απομακρύνονται από την Ευρώπη και θα ήταν σκόπιμο να μην απομακρυνθούμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Να επιστρέψουμε τώρα στους ευρωβουλευτές και στις ευρωβουλευτές ε, βέβαια μεγάλο φάσμα θεμάτων από ζήτημα φορολογίας από την εμπλοκή των προσώπων στην πολιτική η ε, τοποθέτηση του Ιταλού Δημάρχου και βεβαίως και αυτή η τελευταία σας ερώτηση. Κύριε Κάσπαρη, πολλά βέβαια για να απαντήσετε μέσα σε δύο λεπτά. Αυτό που είπατε είναι και από τα βασικά προβλήματα. Πάντα έχουμε μόνο δύο λεπτά. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα εφόσον πρόκειται για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμά εδώ μα απασχολεί πάνω πολύ σε όλε τι κοινοβουλευτικέ, στι περισσότερε κοινοβουλευτικέ ομάδε. Και ένα θέμα το οποίο εξηγεί για ποιο λόγο οι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιημένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ θα είχαμε μεγάλε πλειοψηφίε υπέρ τη επίλυσης του προβλήματο. Όμω, οι χώρες μέλη μας αρνούνται την αρμοδιότητα να λύσουμε το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η φορολογία είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα. Το θέμα αυτό επανέρχεται διαρκώ στην εργασία μου. Οι πολίτε θεωρούν ότι την αρμοδιότητα την έχει δίθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, οι χώρε μέλη δεν μα έχουν δώσει, δεν μα έχουν παραχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή. Οι άνθρωποι όμω τελικώ δεν στρέφονται κατά των κυβερνήσεων του, στρέφονται κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ανένδυμο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί, πρέπει να αλλάξει και πρέπει να γίνει μια συζήτηση που να ξεκαθαρίζει για ποια πράγματα είναι αρμοδιότητα η Ευρώπη και για ποια όχι. Και αυτό νομίζω είναι απαραίτητο να γίνει. Αλλιώ δεν πρόκειται ποτέ να επιλύσουμε τα προβλήματα. Δεύτερο, βοήθεια για τις ε, περιοχέ που έχουν πληγεί από θεομηνίε. Ευτυχώ έχουμε εκεί προγράμματα. Συμφωνώ, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερα. Αλλά είμαστε όμως ειλικρινεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ρυθμίσει τα πάντα. Για πολλά πράγματα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε και με δική μας ευθύνη, στις πατρίδες μας, στις περιφέρειές μας. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι περιμένουμε υπερβολικά πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να υπάρξει παρεξήγηση. Μπορούμε να βοηθήσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να βοηθήσουμε. Όμω η πολιτική και στις χώρες μέλη παίζει σημαντικό ρόλο και οφείλει να δραστηριοποιηθεί και για την πρόληψη των θεομηνιών. Βεβαίω από τη στιγμή που άνθρωποι βρίσκονται σε ανάγκη πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο, βεβαίω είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα για να απαντήσω σε όλα. Γιατί αποστρέφονται τόσο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. ξεφεύγουν, φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το βλέπω, το ζω αυτό. Το πρόβλημα μου όμω είναι όταν κάτι δεν πάει καλά στην χώρα μα, στην πατρίδα μας οι άνθρωποι τότε αντιλαμβάνονται πολύ καλά ποιο κόμμα είναι υπέρ τίνο πράγματο και υπέρ ή κατά άλλου πράγματο. Όμω, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τύπο, τα μίδια λένε πάντα η Ευρώπη. Η Ευρώπη αποφάσισε το ένα, η Ευρώπη αποφάσισε το άλλο. Ποιο όμω στην Ευρώπη ήταν υπέρ και ποιο κατά, δεν το λέει ποτέ κανεί. Ότι εδώ στο κοινοβούλιο συζητούμε, μαλώνουμε, Αυτά δεν τα, τα βλέπουν οι, οι πολίτες και νομίζουν ότι κάπου στην Ευρώπη όλοι κάνουν τα ίδια και γι' αυτό απογοητεύονται και γι' αυτό εκνευρίζονται κατά τη Ευρώπης και λένε θα τους δείξουμε. Και ξεπηδά ο λαϊκισμός. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα λοιπόν για να κατανοήσουν οι πολίτες ποιο κινείται και πώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο αμέσως στην κυρία Σάκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ βεβαίως για όλες τις πολύ ωραία διατυπωμένες ερωτήσεις. Πράγματι πολλά πράγματα τα οποία βρίσκονται μπροστά μας. Φόρο μη δίκαιη φορολόγηση επιχειρήσεων. Αυτά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον έχουμε ωστόσο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Βλέπουμε όμω οι χώρε μέλη, κυβερνήσει των χωρών μελών να ανταγωνίζονται μεταξύ του για να προσελκύσουν τι επιχειρήσει προσφέροντας συχνά πολύ χαμηλούς συντελεστέ φορολογίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις και καμιά φορά μάλιστα και ειδικέ συμφωνίες, special deals. Έχουμε την Επίτροπο Βεστάγκερ που είναι υπεύθυνη για antitrust, για την αντιμετώπιση των trust, εξετάζει τέτοιου συμφωνίε, για παράδειγμα μεταξύ τη μεγάλη εταιρεία Apple και της Ιρλανδία, για να δει μήπω πρόκειται για παράνομη κρατική επιχορήγηση. Χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση. Και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά εκείνα παραδείγματα που μπορούμε να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα εφόσον είμαστε όλοι μαζί. Τώρα, ενθάρρυνση του επιχειρήν. Εγώ είμαι προοδευτική φιλελεύθερη. Θέμα πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μα. Παράδειγμα, διότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Αλλά όταν μιλούμε για ψηφιακή ενιαία αγορά, ακριβώ αυτό προωθούμε τώρα, προσφέρει πολλέ ευκαιρίε και για δημιουργία απασχόληση σε επιχειρήσει ηλεκτρονικών και ηλεκτρονική επεξεργασία. Όμω υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και εκεί για να προωθηθούν αυτέ οι επιχειρήσει να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι του καταναλωτέ σε όλα τα μέρη τη Ευρώπη. χρειάζεται όχι μόνο μια ενιαία αγορά offline αλλά και μια ψηφιακή ενιαία αγορά. Ίσοι κανόνες για όλου. Μιλήσατε και για του σεισμού, που είναι μια από τι καταστροφέ εκείνε που πραγματικά μα έκαναν να αισθανθούμε βαθύτατα και εδώ διότι πρόκειται για θεομηνίες οι οποίες μας συγκλονίζουν και μας. Σα διαβεβαιώνω ότι ο πρόεδρο Ταγιάννη δεν αφήνει να περάσει ούτε μια μέρα χωρί να μα θυμίσει τι συμβαίνει στην Ιταλία. Να είστε απολύτω βέβαιοι λοιπόν ότι το κοιτάζει το θέμα. Νομίζω βέβαια ότι θα χρειαστεί να αρκεστώ σε αυτά. Αλλά επιτρέψτε μου μια σκέψη ακόμα, κυρία Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε περισσότερη ηγεσία, περισσότερη leadership, αλλά και στο επίπεδο των χωρών μελών για να συστρατευτούν οι άνθρωποι και για τα όσα συμβαίνουν εδώ. Το ζήτημα για μένα δεν είναι αν η Ευρώπη κάνει το σωστό ή το λάθο. Γίνεται πιο πολυφωνική και πιο ζωντανή όταν μιλούμε για τη γεωργία, για την ψηφιακή ενιαία αγορά, για την κοινή άμυνα ή για άλλα συγκεκριμένα θέματα. Ολοκληρώνοντα λοιπόν, νομίζω να σταματήσουμε να μιλούμε μοναχά για την Ευρώπη διαρκώ, να αρχίσουμε να συζητούμε πολιτικέ, να κάνουμε πολιτικέ συζητήσει, ποια είναι τα σωστά θέματα και ποιο είναι ο σωστό τρόπο λύση. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε εδώ. Thank you very much, um, to both. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο και όλους όσοι συμμετείχατε στη συζήτηση. Ε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών. Η Βρετανία, όπως ξέρετε, θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ξεκινήσει τη διαδικασία την επόμενη εβδομάδα. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν των 27, Σελίν Κέισμαν, ε, αντιπρόεδρος ε, των νέων ε, Ευρωπαίων από τη Γαλλία, θα θέλαμε να να στρέψει το βλέμμα προς το μέλλον και να δείξει ακριβώς αυτό την Ευρώπη των 27. Κύριε Πρόεδρε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Στις 25 Ιουνίου του 16 πώς αισθανθήκατε. Εγώ αισθάνθηκα λυπημένη για τους φίλους μου, τους ε, Βρετανούς, που θα φύγουν από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εμείς είχαμε ψηφίσει υπέρ της ε, παραμονής της, Ευρω... της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Στη συνέχεια όμως θύμωσα γιατί το παρελθόν επικράτησε επί του, το, του μέλλοντος. Το Brexit είναι ένα hold-up για τους νέους. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ονειρευτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το βλέπουμε και επί επιτόπου. Οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να παρέμβουμε πριν είναι πολύ αργά. Θα πρέπει να δώσουμε ελπίδα, να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δράσει για τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων που εκπροσωπεί και για να επιλύσουμε τις τρέχουσες κρίσεις. Εάν οι ευρωσκεπτικιστές και οι ξενόφοβοι προσπαθούν να διαλύσουν την Ευρώπη, εμείς θα πρέπει να αποτελέσουμε το αντίπαλο δέος. Εδώ και δύο εβδομάδες οι Γάλλοι νέοι έκαναν μία διάσκεψη δύο εβδομάδες πριν καλώντας νέους από όλο τον κόσμο. Και έτσι καταφέραμε να γράψουμε ένα νέο σύνταγμα της Ευρώπης που απαρτίζεται από 12 κεφάλαια. Αυτό δείχνει ότι η δική μας ε, ε, γενιά κάνει προτάσεις επικοδομητικές για το μέλλον της Ευρώπης. Θέλουμε μια πιο δημοκρατική Ευρώπη και πιο ενωμένη. Αυτό δείχνει ότι θέλουμε μια νέα Ευρώπη καινοτόμη που να ανταποκρίνεται στο ιδρυτικό της πνεύμα. Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε, την οποία όμως δεν επιβάλλουμε. Thank you. σας ευχαριστώ πολύ. Ευρωβουλευτές. Πρώτος ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από τους πολίτες της και στη σήμερα υπάρχει κάποιο πρόβλημα μικροφώνου. Ίσως να διορθωθεί τώρα. Ευχαριστώ λοιπόν έλεγα κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πολίτε τη και οι ευκαιρίε όπω η σημερινή έχουν τεράστια σημασία. Θα πρέπει να συναποφασίσουμε το μέλλον μα. Ο βρετανικό λαό αποφάσισε να καταλήψει την Ευρώπη από τι μεγαλύτερε προκλήσει από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμω γεγονό και δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα στι επιθυμίε μα. Το αντίθετο συμβαίνει. Όμως είναι μια πρόκληση που μπορεί να γίνει ευκαιρία. Εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους οι Βρετανοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον τρόπο που λειτουργεί. Έχουμε το καθήκον να το αντιμετωπίσουμε. Το ευρωπαϊκό project δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όμως τώρα το υπόδειγμα λιτότητας το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί τον κόσμο σε φτώχεια. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί και εφαρμόζει ε, πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε βάθεμα των ανισοτήτων. Χωρίς αλλαγή, χωρίς τροποποίηση των συνθήκων δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανέλθει στον δρόμο της εξυπηρέτησης των πολιτών της. Χρειάζεται ανάπτυξη μιας κοινωνικής και δίκαιης Ευρώπη για να εξυπηρετήσει τους στόχους της πλήρους απασχόλησης. Και αυτά τα λέει και η συνθήκη μαζί με τις οριζόντιες κοινωνικές ρήτρες και με την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η λευκή βίβλος ε, του Jean-Claude Juncker πρέπει να πάει ένα σφάλμα. Δεν επιφέρει αναθεώρηση στα βασικά κείμενα, στις συνθήκες. Το Brexit μπορεί να σημάνει ωστόσο το πρώτο κομματάκι του εφέ του ντόμινο ο κόσμος γνωρίζει ότι έχει ηθικό και ιστορικό καθήκον να κάνουν ό,τι μπορούν όλοι ώστε να αποφευθεί αυτό το ντόμινο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Δεν είπα ότι ο κύριος Καστάλντο είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της ε, Ελευθερίας και Δημοκρατίας, Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και κρατώ το μήνυμα που προαναφέρατε. Κατά τη διάσκεψη των νέων στην ε, πατρίδα σας. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά για να σας πω ότι ερχόσαστε με το σωστό μήνα για, μήνυμα συγγνώμη, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα που θα πρέπει να προσυπογράψουμε στη Ρώμη όταν θα συναντηθούμε για την πανηγυρική αυτή υπογραφή. Μιλάμε για ειρήνη και ευημερία. Αυτό είναι το διακύβευμα, αλλά και το δικαίωμά μας στην ευτυχία. Οι νέοι στην Ευρώπη είναι αυτοί που θα πρέπει να προβάλλουν αυτό το μήνυμα. Στη Ρώμη, 60 χρόνια μετά, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μία αγορά και μόνο. Θα πρέπει να είμαστε μία πλήρης πολιτική ε, οντότητα με την ε, πολιτισμική και κοινωνική της πτυχή, καθώς και την οικονομική. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να είναι πραγματικά πολίτες. Και αυτό είναι το μεγάλο σας μήνυμα. Και θα πρέπει να προβάλλετε και επιχειρήματα για να πείσετε τους άλλους. Γιατί χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Γιατί αν παραμείνουμε μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, την ψηφιακή επανάσταση, έτσι όλοι, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και προστασία και η Ευρώπη θα τα καταφέρει ώστε να έχετε εσείς ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι αυτή είναι η φωνή σας που θα πρέπει να διατρανωθεί και στη Ρώμη. Αλλά σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ. Εντάξει, είδα τους αριθμούς, δεν χρειάζεται να τους κρατάτε. Ε, σε αυτό το θέμα υπήρχε μεγάλο ε, ενδιαφέρον. Το 690 έχει το λόγο. Είμαι ο Γιούλιαν Σούλτ, έρχομαι από τη Γερμανία, είμαι 17 χρονών και φέτο ε, θα ψηφίσω για πρώτη φορά στη Γερμανία. Ε, και νομίζω όσοι βρίσκονται στην αίθουσα θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι η δική μου γενιά είναι εκείνη που πρέπει να στηρίξει την Ευρώπη, ε, είναι υπεύθυνη για το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, πείσουμε τους ε, συνομιλίκους μας ε, να συμμετέχουν και αυτοί να αποφασίσουν γιατί μόνο έτσι θα υπάρχουν εγγυήσει ε, για το μέλλον της πολιτικής. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στη δική μου γενιά, μειώνεται το ενδιαφέρον. Και το είδαμε και με την ψηφοφορία για το Brexit. Πολλοί δεν πήγαν καν να ψηφίσουν, πολλοί νέοι. Αυτό πρέπει να εμποδιστεί στο μέλλον. Οι νέοι πρέπει να ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, γενικά για την πολιτική και τελειώνοντας θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να μεριμνήσει έτσι ώστε για τους νέους ε, να υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον για την πολιτική. Και τώρα η 3.21 παρακαλώ, ερώτηση. 3.21. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ποια είστε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Αν που είμαι μέλος του Students for Europe. Είμαι φοιτήτρια στο Μάστριχτ. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Θα πρέπει όμως να φτάσουμε σε συγκεκριμένα ευεργετήματα. Δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι ελευθερίες που προασπίζονται. Δεν θα πρέπει ε, ε, να είμαστε μία αποσπασμένη οντότητα. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για να αντιμετωπίσουμε τα υπαρξιακά μας ερωτήματα. Πώς θα σπάσει η φούσκα μέσα στην οποία είναι κρυμμένοι τα πολιτικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, πολύ και η φωτογραφία αυτή, το πανό αυτό ήταν πολύ καλό. 809. 809 τώρα, νομίζω ότι είναι πίσω-πίσω στην αίθουσα. Λέγομαι Λάουρα Χιν από το Ούρζεν, Γερμανία. Εδώ βλέπω στην ημερήσια διάταξή σας ότι πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον να βρούμε λύσεις με κοινή προσπάθεια. Εμένα με ενδιαφέρει το προσφυγικό. Εκεί χρειάζονται καλύτερες λύσεις. Και ιδίως ό,τι αφορά μια ενωμένη στάση. Γιατί χώρες όπως η Πολωνία δεν υποδέχεται καθόλου πρόσφυγες. Θεωρώ ότι εμείς οι Γερμανοί υποδεχτήκαμε πάρα πολλούς πρόσφυγες. Και η Άγγελα Μέρκελ έπαιξε υποδειγματικό ρόλο. Νομίζω όμω ότι χρειάζεται ενωμένη στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για να υπάρξει αυτή πρέπει και χώρε όπω η Πολωνία να δηλώσουν ότι είναι διατεθειμένε να υποδεχτούν πρόσφυγε. Αυτό ήθελα να πω. Τελευταίο, Τελευταίος, η τελευταία, 609, 609, 609. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Σόνια Φανάσελ από τους νέους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές. Ορισμένοι επιδοκίμασαν το Brexit, ότι δηλαδή επιτέλους θα προχωρήσει η Ευρώπη και θα γίνει πιο συμπεριληπτική, αφήνοντας κάποιους απ' έξω. Αυτό όμως είναι αμφισβητήσιμο. Ορισμένες φορές το αίσθημα που μας διακατέχει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνεται κυρίως στην οικονομική ολοκλήρωση, αφήνοντας απ' έξω άλλα θέματα. Για παράδειγμα, εμείς λησμονούμε ότι η Ευρώπη μας είναι πρώτα-πρώτα ένα πολιτικό έργο ολοκλήρωσης. Ειρήνη, ευημερία, αλληλεγγύη. Πώς θα κάνουμε πιο ισχυρή την Ένωση, ακόμα και αν παραμείνει μονάχα Ένωση των 27. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ επίσης, λέει η πρόεδρος κυρία Μαρκίνες. Οι δύο ε, συναδελφοί μου τώρα, εσείς πρώτα κυρία Ροντρίγκες, αν θέλετε απαντήστε πώς να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω στη γενική συζήτηση που κάναμε. Πώς μπορούμε δηλαδή να προκαλέσουμε πάλι το ενδιαφέρον για την Ευρώπη, την επιθυμία να συμμετάσχουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Να σας πω κάτι από τη δική μου προσωπική ιστορία άρχισα με μια ε, εμπειρία προ-έρασμος, πριν από τον έρασμο. Με συνεργασία με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο και αυτό άλλαξε σε βάθος τη ζωή μου. Είμαι βεβαία ότι όλες και όλοι σας έχετε τέτοιου είδους εμπειρίες και αυτή τη στιγμή έχετε αυτή την εμπειρία. Σίγουρα αυτό άλλαξε τη ζωή σας. Η απάντησή μου λοιπόν στην ερώτησή σας είναι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες εμπειρίες κοινέ συνεργασίας σε όλα τα μέτωπα. Όταν μαθαίνουμε, όταν διδασκόμαστε, όταν ε, πιάνουμε την πρώτη μας δουλειά, όταν ε, μετακινούμεθα σε μια νέα ευρωπαϊκή πόλη και κάνουμε φίλες και φίλους εκεί, όταν συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε κάτι το νέο στις τέχνες, στην επιστήμη, όταν συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε ανθρωπιστικά προβλήματα. Δεν μπορώ να λησμονήσω όταν αρχίσαμε να έχουμε το αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης που είδαμε πολύ ζωντανού νέους Ευρωπαίους, νέους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονταν για πραγματική ανταπόκριση στο πρόβλημα του προσφυγικού. Όταν έχουμε τρίτες χώρες σε όλο τον κόσμο, πάμε να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και να έχουν και αυτοί ευκαιρία στη ζωή τους. Σε όλα αυτά, οι Ευρωπαίες νέοι, οι Ευρωπαίες νέες και νέοι μπορούν να συνεργαστούν και μπορούν έτσι να μεταφέρουν αυτή την επιθυμία συμμετοχή στην Ευρώπη και σε όλες τις άλλες ηλικίε. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε εμπειρία ενός νέου είδους δημοκρατίας. Και αυτό πρέπει να είναι το υπόδειγμα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εσείς κύριε Καστάλτο. Madame Chair, je vais répondre euh, avec quelques mots. Θα απαντήσω στα γαλλικά γιατί και εγώ είμαι παιδί της ε, γενιάς του μου. Δύο χρόνια πέρασα στη Γαλλία και τώρα θα μιλήσω Ιταλικά. Θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Φυσικά θα πρέπει να συμμετέχουν οι νέοι και αυτό σημαίνει μία συμμετοχική προσέγγιση. Θα πρέπει να βασιστούμε στην άμεση συμμετοχή, στην συμμετοχική δημοκρατία. Μία έκθεση που ψηφίσαμε λίγο πριν, γιατί με μικρά βήματα μπορούμε να φτάσουμε σε μία πολιτική συνείδηση. Και πιστεύω ότι η πρωτοβουλία Ευρώπη για τους πολίτες θα πρέπει να αποτελέσει ένα πραγματικό μέσο και να μην μας παρεμποδίσει η Κομισιόν. Πώς μπορούμε να διαδώσουμε καλύτερα τις ελευθερίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάζουμε τον πύχη λίγο πιο ψηλά. Η κοινωνική Ευρώπη είναι η μεγάλη ξεχασμένη γιατί δεν την θέλησαν πολύ. Οι συνθήκες τώρα μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε πιο μακριά. Δεν αρκεί να το λέμε, να μείνουμε στα λόγια και μόνο, αλλά να θέσουμε τα μέσα για να εφαρμόσουμε αυτή την ολοκλήρωση και όχι το αντίθετο, δηλαδή να κάνουμε την ολοκλήρωση μέσω λιτότητας. Ως προς την αλληλεγγύη μιλήσαμε για κοινέ λύσεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Μερικές ε, χώρες δεν δέχτηκαν αυτές τις αποφάσεις. Υπήρχαν ε, διπλά μέτρα και σταθμά, το οποίο ήταν λανθασμένο. Θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις από όλους, αλλιώς δεν θα πάμε μακριά περνάει ο χρόνος ή θα συνεχίσουμε την ιστορία της Ευρώπης ή θα την παρεμποδίσουμε φτάνοντας σε μηδενικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ σε όλους που συμμετείχαν. Τώρα, η ασφάλεια και η προσθέσια των πολιτών σε ταραχώδεις καιρούς. Ξέρετε ότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες σε θέματα ασφάλειας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πάζρα, ο οποίος εργάζεται στο King's College στο Λονδίνο, στο κέντρο κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Ένα χρόνο πριν οι τρομοκρατικές ενέργειες της 22 Μαρτίου στις Βρυξέλλες μας ε, έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος. Οι αδελφοί Ελμπακράουι έχουν, είχαν μια μακρά ιστορία με τη βία. Παρέμειναν στις φυλακές, εκεί ε, ασχολήθηκαν και προσιλητίστηκαν στο τζιχάτ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές ε, οι εξτραμεστικές τάσεις στην ουσία διονγκούνται και γνωρίζουμε ότι αυτοί που ταξίδεψαν στη Συρία είναι αυτοί που είχαν και εγκληματικό ποινικό μητρό. Δυστυχώς στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης είχαν ανάμιξη με το έγκλημα και έχουν αντιφατική συμπεριφορά. Πολλούν ναρκωτικά ή τα χρησιμοποιούν και αυτό το είδαμε και στο ε, Βερολίνο αλλά και στο αεροδρόμιο του Ορλή. Άρα είναι δύσκολο να υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ εγκλήματος και τρομοκρατίας. Οι προτάσεις για το πώς θα πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη δείχνουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, κοινή βάση χρησιμοποίησης των πληροφοριών και ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για να είναι ε, αποτελεσματική συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν τα δίκτυα καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Ευρώπη για να γνωρίσουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην τομοκρατία. Εάν ε, μου έλεγαν ε, ότι θα είχαμε πολλούς ομιλητές, πολλούς ερωτώντες τελευταία ε, στο τελευταίο θέμα θα, θα το πίστευα και πράγματι ε, έτσι είναι. Θα αναγκαστώ μερικούς να μην τους δώσω το λόγο. η κυρία Μετσόλο, με συγχωρείτε, ναι, από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όσοι πιστεύουν ότι είμαστε εδώ μακριά από το σπίτι μας ποτέ θα ξεχάσουν αυτό το αίσθημα φόβου, αγωνίας, ε, αγανάκτησης ε, για τα θύματα της τρομοκτικής επίθεσης πριν από ένα χρόνο. Όμως ε, αυτό το σοκ έδωσε τη θέση του σε μία λύπη και το γεγονό, το συνέστημα ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα αίτια και την ρίζοσπαστικοποίηση που μαστίζει την κοινωνία μας. Αν ρωτήσω τους συμπολίτες μας τι τους είναι πιο σημαντικό, η δική τους απάντηση απάντηση είναι ότι θα ήθελαν να απολαμβάνουν το βασικό δικαίωμα που είναι να αισθάνονται ασφαλείς ε, ε, σε όλα αυτά που κάνουν, να ζουν τη ζωή που επιλέγουν να ζουν. Σε αυτό λοιπόν εδώ το Κοινοβούλιο δουλέψαμε σκληρά, πρώτα απ' όλα για να επιταχύνουμε τις προσπάθειες ώστε να υπάρχουν κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες για καλύτερη ενημέρωση των ε, πολιτών που ταξιδεύουν από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύστημα PNR. Έχουμε πιέσει λοιπόν για στρατηγικές κατά της παστικοποίηση, ε, διώκουμε του ανθρώπου που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, καταζητούμε το χρήμα και ψάχνουμε να βρούμε δρόμου για να στηρίξουμε τα θύματα τη τρομοκρατία. Διότι η τρομοκρατία έχει πάρα πολλά ε, κρυφά ε, θύματα που στιγματίζουν πολλέ γενιέ. Θέλουμε αυτοί να αποκτήσουν φωνή, να του στηρίξουμε να επανέλθουν στη ζωή και να μην ξεχνάμε όλου αυτού που χάσαμε. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που κάναμε, όμω όλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλέψουμε περισσότερο στην ανταλλαγή των πληροφοριών, να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματά μας της πληροφορικής λειτουργούν άψογα και σε συνδυασμό, διότι η πρόληψη και η δίωξη της ε, εγκληματικής συμπεριφοράς ε, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό μητρό που να λειτουργεί. Να βελτιώσουμε τη χρήση των βιομετρικών ε, δεδομένων. Από τα κενά στο Βερολίνο είδαμε ανθρώπους που είχαν 40 διαφορετικέ πολιτικές ταυτότητες. Η τρομοκρατία είναι μια παγκόσμια απειλή που απαιτεί και μια παγκόσμια απάντηση στην εργασία με τρίτες χώρες γιατί ε, είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε τελικά να καταφέρουμε και να επιτύχουμε το στόχο μας. And now I invite Monica of the European... Η Μόνικα Μάκοβε από την ομάδα ε, Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ απευθύνω χαιρετισμό προ όλε και όλου. Θα απαντήσω πρώτα στην ερώτηση του Ράιαν για τη συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ χωρών μερών σε ό,τι αφορά την ε, ε, γνωστοποίηση πληροφοριών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο λείπει. Και αυτό οδήγησε σε αυτέ τι ατυχεί τρομοκρατικές επιθέσεις. Τώρα ευτυχώ έχουμε περισσότερε τράπεζε δεδομένων. Έχουμε τράπεζα δεδομένων για τι προξενικέ θεωρήσει, έχουμε το σύστημα πληροφοριών Schengen, και άλλε τράπεζε δεδομένων. Ε, Βεβαίω η Ευρωπόλ έχει επίση τη δική τη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτέ οι τράπεζε δεδομένων μέχρι τι επιθέσει αυτέ, δηλαδή μέχρι πριν από ένα χρόνο στην ουσία, ήταν α πούμε μισοάδιες, διότι οι χώρες μέλη δεν ε, θεωρούσαν αναγκαίο να τι γεμίζουν με δεδομένα. Υπήρχε η τάση των χωρών μελών να κρατάνε τι πληροφορίε για τον εαυτό του. Δεν θέλουν δηλαδή να μοιράζονται τις προφορίες που συλλέγουν οι υπηρεσίε του με άλλε χώρε μέλη είτε διότι δεν εμπιστεύονται τις άλλες χώρες μέλη για άλλους λόγους. Αυτό πρέπει να αλλάξει και έχει αρχίσει να αλλάζει. Για παράδειγμα η Ευρωπόλ που είναι ευρωπαϊκός οργανισμός έλαβε πληροφορίες από χώρες μέλη με 8 εκατομμύρια νέα πληροφοριακά στοιχεία μέχρι πρόσφατα, μέσα σε ένα χρόνο. Όλες οι χώρες μέλη καλούνται τώρα να πληρώνουν τις τράπεζες δεδομένων με ακριβή δεδομένα και μάλιστα ταχύτατα. Αυτή η συνεργασία έχει τη δυνατότητα να σταματήσει άτομα τα οποία έχουν τρομοκρατικές ή εγκληματικές προθέσεις. Να τους εμποδίσει να μεταβαίνουν από τη Γερμανία στη Γαλλία, στο Βέλγιο ή να μπουν καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάνε στη Συρία και να επανέλθουν με διαφορετική ταυτότητα για παράδειγμα, γιατί και αυτό ήταν δυνατό. Εργαζόμαστε και πάνω στη συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων, σε ε, εικόνες του προσώπου και στους άλλους ελέγχους που διεξάγονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο μέλλον, επειδή οι εμπειρογνώμονες λένε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν είναι πλέον ο πιο ασφαλής τρόπος για να ταυτοποιηθεί κάποιο, γιατί μπορούν και αλλάζουν ή τα καταστρέφουν τα δακτυλικά αποτυπώματα στα δακτυλά του. Θεωρούμε ότι το επόμενο θα πρέπει να είναι η, αυτό το fingerprint τη κόρη του ματιού, τη ήρυδα του ματιού. Λέω λοιπόν ότι η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Θα πρέπει να το αντιληφθούν οι χώρε αυτέ μέλη. Να το αντιληφθούμε όλοι. Εδώ στο Κοινοβούλιο συμμετέχουμε ευρωβουλευτέ από πολλέ, από όλε τι χώρε. Πρέπει να συνεργαστούμε. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπηρεσίε συλλογή προφοριών σε όλε τι χώρε μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, λέει η Πρόεδρο. Μόνο τέσσερι. Και ζητώ συγγνώμη από πριν. από πριν. Το νούμερο τρία. Λέγομαι Βέρελ από τη Γερμανία. Αλλάζουν οι καιροί. Νέε απειλέ που μας αναγκάζουν να λαμβάνουμε νέα μέτρα. Ε, ακούστηκαν ήδη πολλά νέα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια των πολιτών. Ωστόσο, να μην, ε- να μην υπερβάλλουμε κιόλας, διότι όποιος τελικά θυσιάζει την ελευθερία στο βωμό της ε, ασφάλειας, χάνει τελικά και τα δύο. Θα χρειαστεί να δοθούν νομοθετικά επαρκή δικαιώματα στις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά Ξαναλέω, χωρίς υπερβολέ. Όχι επειδή έγινε τώρα μια τρομοκρατική επίθεση να περικοπούν τα δικαιώματα των πολιτών. Ασφαλώς, του ύψου το αγαθό είναι η ασφάλεια. Αλλά, επαναλαμβάνω, όχι ε, σε βάρος της ελευθερίας. 245. Είμαι ο Αντώνιο Κοέλιο Προέρχομαι από την Πορτογαλία. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφραστώ εξ ονόματος της Πορτογαλίας και ιδιαίτερα της Βόρειας Πορτογαλίας. Προέρχομαι από μια περιοχή που είναι πολύ φτωχή. Λυπάμαι ιδιαίτερα διότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν πάντα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε ε, επιθέσεις και ε, οι επιθέσεις αυτές αφορούν αγρότες, πολίτες, ε, τοπικούς φορείς και ούτω καθεξής. Δυστυχώς στον αγροτικό κόσμο υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τις περιφέρειες που έχουν απεριμωθεί. Δυστυχώς δεν μπορείτε να κατανοήσετε αυτό το ζήτημα γιατί σήμερα ο αγροτικός κόσμος, ο φτωχός αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απομόνωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς που προωθούμε θέματα βιοπικιλότητας, προωθούμε και τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης περιοχής. 571 571 έχετε το λόγο. Είμαι από το Δημοκρατικό ε, Κόμμα του Βελγίου και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ε, έχουμε κάνει και πρέπει να γίνουν πολλές επενδύσεις στον τομέα της ε, πληροφορικής έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Νομίζω ότι δεν ε, αρκούν τα εργαλεία πληροφορικής που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να έχουμε κατά νου και εκείνους ε, που στιγματίζονται αδιάκοπα και θεωρούνται υπεύθυνοι για την τρομοκρατία. Αναφέρομαι στους πολίτες από τη Βόρεια Αφρική. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα του οίκου μας. Ας ε, προσπαθήσουμε να εμφανιζόμαστε με λιγότερα αισθήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Θα ήθελα λοιπόν να ε, παραθέσω και κάτι που είπε ο πρόεδρος ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Βρυξέλλες στιγματίστηκαν και συνδέονται με την τρομοκρατία. Άρα δηλαδή να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, να αρχίσουμε τα του οίκου μας και να είμαστε λιγότερο ρατσιστές με λιγότερα συναισθήματα ξενοφοβίας. ξενοφοβής. 1-4-8 παρακαλώ. Το ένα, 4 8 Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ε, έρχομαι από την Δανία και πρέπει να σας πω, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι πράγματι χρειαζόμαστε την ε, ευρωπαϊκή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεις. Πρέπει να μαθαίνουμε από ε, τα μαθήματα που παίρνουμε από άλλους θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία της σημερινής ε, συνάντησης να θέσω το εξής ερώτημα. Πώς μπορούμε να ε, σταματήσουμε τον καλύτερο τρόπο την τρομοκρατία. Νομίζω η απάντηση προκύπτει από την ίδια τη λέξη τρομοκρατία. Δεν πρέπει να τρομοκρατούμεθα. Δεν πρέπει λόγω αυτών των ε, ελεηνών πράξεων να αποεμπολίσουμε τα ατομικά μας δικαιώματα. Όλο και περισσότεροι αυτό οι πολίτες παρακολουθούνται. Εγώ όμως βέβαια δεν συμφωνώ με το να υπάρχει υπερβολική παρακολούθηση. Και πολύ καλό το γεγονός ότι θεσπίστηκε και σχετική οδηγία επ' αυτού. Υπάρχει και ένας νέος νόμος που αναφέρεται στα στοιχεία που αφορούν στις επιχειρήσεις και ε, μπορεί κανείς ε, να επιθυμεί οι υπηρεσίες ασφαλείας, ε, αντικατασκοπίας να δουλεύουν στοχευμένα. Οφείλουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών σε όλη την υπηρό μας. Νομίζω ότι, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να απεμπολούμε τις αρχές μας, ε, γι' αυτό υπάρχουν αρχές, ε, για τις δύσκολες καταστάσεις όταν τα πράγματα είναι άβολα. Ευχαριστώ και ας επιστρέψουμε τώρα στις κυρίες Μετσόλα και Μακοβέ Πρώτα κυρία Μετσόλα θα τηρήσω όμως αυστηρά το όριο χρόνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχει μιλήσει κανείς ακόμα την μητρική μου γλώσσα, τα Μαλτέζικα, γι' αυτό θα το κάνω εγώ και θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλες και όλους που έθεσαν ερωτήσεις ε, στην διάρκεια της συζητήσεως αυτή. Σύμφωνο με το πρώτο ερώτημα ότι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε διότι εάν πρόκειται να περιορίσουμε τις ελευθερίες που είναι αποτέλεσμα τόσο σκληρών αγώνων εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει ότι τελικά κερδίζουν το παιχνίδι οι τρομοκράτες. Αυτό για μένα εγώ έχω αγωνιστεί και έχω αγωνιστεί πολιτικά για να μπει η χώρα μου η Μάλτα στην, ε, στον χώρο Σέγγεν. Θα χρειαστεί όμως τότε να αντιστρέψουμε όλα αυτά. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αγωνιστούμε περισσότερο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Χρειάζεται βεβαίως να υπερασπιστούμε του, όλους τους πάντες, αυτούς που ζουν στις ε, πόλεις, αυτούς που ζουν στα χωριά. Είμαι μητέρα. Τα παιδιά μου με ρωτούν γιατί όταν πηγαίνω στο σχολείο ή όταν βγαίνω έξω βλέπω παντού στρατιώτες. Και όταν συγκρίνω τη ζωή των παιδιών μου με τη ζωή που έζησα εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, βλέπω ότι η δική τους ζωή τώρα γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Είναι και πολύ πιο δύσκολο για μένα να έχω τα παιδιά μου ασφαλή από ό,τι ήταν για τους γονείς μου να έχουν εμένα ασφαλή για τα δεδομένα. Για τα δεδομένα πρέπει να κάνουμε πράγματι πολύ περισσότερα. Εάν δώσουμε στις αρχές επιβολής του νόμου, αστυνομικές και άλλες, περισσότερες αρμοδιότητες για να ανταλλάσσουν πληροφορίες, δεδομένα, μπορούμε τότε να προλάβουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. για να μην είμαστε υποχρεωμένες και υποχρεωμένοι να επανερχόμαστε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλούμε ξανά για τέτοιες τραγικές υποθέσεις. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Αυτό μπορώ να σας υποσχεθώ. Χρειάζεται βεβαίω να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία. Η κυρία Μακοβέη, πάλι βεβαίω προσοχή στο χρόνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ακολουθήσω το πρόγραμμα ε, συγγνώμη, το, το υπόδειγμα της ε, Ρομπέρτα και θα μιλήσω ρουμανικά. Εγώ αυτή τη φορά ελπίζω να υπάρχουν και Ρουμάνοι μέσα στην αίθουσα. Υπάρχουν Ρουμάνοι ή Ρουμάνες μέσα στην αίθουσα? Α, ωραία. Μπράβο λοιπόν. Ε, να, συνεχίζω τότε στα ρουμανικά. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ελευθερίες των πολιτών όταν μιλάμε για μία εξισορρόπηση ελευθεριών και ασφάλειας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μία σωστή ποιότητα ζωής. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε κατά της ιδιωτικής ζωής. Όμως όταν υπάρχουν υπάρχουν στοιχεία ως προς ποινικά μητρώα, δακτυλικά αποτυπώματα και ούτω καθεξής. Το κακό είναι ότι δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών και γι' αυτό έγιναν και οι επιθέσεις, γιατί δεν ήμασταν συντονισμένοι. Μιλάμε για συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν οι πληροφορίες Άρα θα πρέπει να συντονιστούμε και να υπάρχει διαφάνεια. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί διοκτήτες επιχειρήσεων για να μην ξεπλένεται ε, βρωμικό χρήμα μέσω των επιχειρήσεων. Να μην γίνεται χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας από μεγάλες επιχειρήσεις. Να υπάρχει διαφάνεια γιατί οι φορολογούμενοι καταβάλουν το τίμημα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, προωθήσουμε την πίστη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, γνωρίζουμε ότι το τίμημα είναι πολύ υψηλό και δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι είμαστε ίσοι. Ε, ελπίζω οι επισκέπτες να μην ε, με φοβούνται όταν χτυπάω το σφυράκι μου. Είμαι υποχρεωμένη. Τώρα περνάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους τις κλιματικές ή κλιματικές αλλαγές και η προστασία του πλανήτη μας. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την Μάγδα Στόκλιεβιτς που είναι διευθύντρια του οργανισμού Friends of the Earth Europe να μας μιλήσει. Μιλάμε για μια κατεπίγουσα ανάγκη. Οι κλιματικές αλλαγές συμβαίνουν και είναι πραγματική απειλή. Δεν είναι φάρσα αλλάζουν τα πράγματα παγκοσμίως. Θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς Κελσίου και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μην έχουμε αύξηση θερμοκρασίας πάνω από 1,5 βαθμό το ε, σύστημα ενέργειας της Ευρώπης μέχρι το 2020 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα. Γι' αυτό θα πρέπει να μην έχουμε πια εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να έχουμε ένα μέλλον ελεύθερο από τα καύσιμα αυτά. Να μην ε, λοιπόν χρηματοδοτούμε το, το πετρέλαιο και τα υποπαράγωγά του. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μας σύστημα και η οικονομία μας να γίνει πραγματικά κυκλική οικονομία. Οι πολίτες είναι στο προσκήνιο αυτής της αλλαγής, συμμετέχουν σε οργανώσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει τέτοια εξάρτηση πλέον από τα ορυκτά καύσιμα. Να υπάρχει σωστή μετάβαση και κανένας να μην μείνει πίσω. Ε, χαίρομαι που είμαι Πολωνή, αλλά ντρέπομαι για αυτά που κάνει η πολωνική κυβέρνηση ως προς την ενέργεια και το κλίμα όλοι οι κυβερνήτες είναι υπόλογοι. Τι κάνουν οι πολιτικοί στις χώρες σας. Θα πρέπει να υποβάλουμε ερωτήματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ενεργειακό πακέτο θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο όταν βγει και ψηφιστεί από το σώμα σας σε σχέση με το αρχικό που υποβλήθηκε. Και τώρα λοιπόν, ε, για να δούμε λιγάκι την αντίδραση των ε, ευρωβουλευτών, ο κύριος Εκχάτ εκ μέρους ε, των Πρεσίων παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Νομίζω είναι πολύ ωραίο το ότι βλέπουμε για 60 χρόνια έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να διεξάγουμε αυτές τις συζητήσεις. Αισθάνομαι όμως ότι διαπιστώνεται υπάρχουν κάποια προβλήματα. Γιατί αν ακούς κανείς αυτά που ελέγχθησαν σήμερα εδώ φαίνεται ότι όλοι συμφωνούν. Προσέξτε όμως, ε, δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνούμε σε αυτό το θεσμό έχουμε έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι πολύ καλό το ότι είμαστε ένας δημοκρατικός θεσμός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσά μας. Όταν ακούει ε, κανείς να μιλάνε μερικοί για φοροαποφυγή, άλλοι λένε όχι είναι φορολογικός ανταγωνισμός ή θεμητό εμπόριο. Όλοι το λένε, αλλά εσείς πρέπει να ρωτήσετε έναν πολιτικό γιατί οι εταιρείε δεν μπορούν μπορούν να ενάγουν τις κυβερνήσεις τους. Τέτοιου είδους θέματα πρέπει να συζητούνται. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέλουν οι εταιρείε να μπορούν να ε, ενάγουν, όπως είπαμε, τις κυβερνήσεις τους. Τέτοιου είδους θέματα πρέπει να συζητούνται. Και το ίδιο ισχύει και για την ε, κλιματική αλλαγή. Όλοι λένε πόσο σημαντικό ήταν το Παρίσι, η Συμφωνία του Παρισιού, πόσο θεμελιώδου σημασίες, αλλά πρέπει να τους ρωτήσετε και τι θα αλλάξετε, τι θα μεταφερθεί στην πολιτική για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Εγώ έρχομαι στην Ολλανδία. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εκλογέ και μόνο τρία κόμματα εφαρμόζουν αυτά που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι. Ακόμα και οι σοσιαλδημοκράτε. Συγγνώμη, Τζο, που κάθισε δίπλα μου, και αυτοί δεν έκαναν αρκετά για να εφαρμοστεί η συμφωνία του Παρισιού. Και αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Εντάξει, πολύ ωραίο που έχουμε 60 χρόνια δημοκρατία, αλλά να μην ακούσουμε ακούτε μόνο ωραία λόγια από τους πολιτικούς σας, να διασφαλίσετε και ότι οι πολιτικοί θα μεταφέρουν όλα αυτά στην πράξη. Πολύ ωραία. Ε, θα πάρετε το βραβείο του Ευρωβουλευτή που τήρησε ακριβώς το χρόνο του. Είχαμε λοιπόν ήδη την εισαγωγή. Κύριε Λάνελ έχετε το λόγο. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος ε, και είμαι χαρούμενος που είσαστε όλοι εδώ γιατί είμαι και πρόεδρος ε, του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Κινήματος. Ελπίζω να έχουμε ένα νέο ευρωπαϊκό κίνημα για τα 60 χρόνια από τη συνθήκη της Ρώμης γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιαχτεί για του πολίτε, όχι για τι κυβερνήσει. Όλοι κοιτάνε τι γίνεται στο Στρασβούργο, στι Βρυξέλλε. κανεί όμω δεν δραστηριοποιείται και χαίρομαι πάρα πολύ που τι προηγούμενε εβδομάδε χιλιάδε ανθρώπων κατέβηκαν στου δρόμους, στι πλατείε και στη Ρώμη το επόμενο Σάββατο θα έχουμε δεκάδες χιλιάδε που θα κάνουν πορεία για την Ευρώπη. Για μια Ευρώπη που προσφέρει ελπίδα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια μια Ευρώπη που υπάρχει για το μέλλον και χαράσει τις πολιτικές που χρειαζόμαστε κατά τον 21ο αιώνα. Εγώ ασχολούμαι πάρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ε, περιβαλλοντική προστασία πριν καν ιδρυθεί το κόμμα των Πρασίνων. Και ε, εντάξει, παρόλα αυτά θεωρώ ότι συνεργαζόμαστε η εκβιομηχάνηση ξεκίνησε στην Ευρώπη πριν από 250 χρόνια. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να είμαστε ηγέτες στον κόσμο. Είμαι και επικεφαλής της αντιπροσωπείας με την Κίνα. Βλέπουμε τι κάνει η Κίνα. Κάνει άλματα. Άρα δηλαδή θα πρέπει και εμείς ε, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ε, όχι μόνο για να ε, με λόγια να τα στρώμεθα υπέρ της οικολογίας αλλά να προβαίνουμε και σε πράξεις. Η Κίνα αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί σε 10 βασικούς τομείς, να ε, διεκδικήσει την καλύτερη τεχνολογία, ηλεκτρικά, ε, αυτοκίνητα, ρομποτική, που μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για οικονομική, και κοινωνική πρόοδο, αλλά όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, πρώτα να σώσουμε τον πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ χωρίς πολλά λόγια. Αριθμός 76. Παρακαλώ, ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Έρχομαι από την Ιαλική Λιόν. Ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι η κλιματική κρίση είναι στην ουσία η μητέρα όλων των κρίσεων θα έλεγα. Ωστόσο, εδώ και λίγο χρόνο μόλις οι Ευρωπαίοι βουλευτές επικύρωσαν την Συμφωνία Εμπορικών Συναλλαγών με τον Καναδά και που σημαίνει ακόμα περισσότερο διοξείδιο του άνθρακου στην ατμόσφαιρα εν τέλει. Εδώ βλέπω κάποια συμβατότητα ανάμεσα στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί το 2015 μόλις στο Παρίσι στην ε, διάσκεψη για το κλίμα και σε αυτό το αποτέλεσμα των ελεύθερων συναλλαγών με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η συμφωνία αυτή. Θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες σας. 250. Αριθμός 250. Ορίστε. Ονομάζομαι Ρικάρντο Ινκαρνασάου, προέρχομαι από την ε, Πορτογαλία. Αυτό το θέμα του περιβάλλοντος είναι άκρος σημαντικό. Στην ουσία προσπαθούμε να εξεύρουμε λύσεις με λανθασμένες προσεγγίσεις. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πραγματικά τις κλιματικές αλλαγές. Στις αρχές της ε, ε, δεκαετίας το 90 ή το 2000 ε, δεν αντιμετωπίσαμε το ζήτημα όπως θα έπρεπε. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πρόσφυγες για περιβαλλοντικούς λόγους οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα τους ακριβώς γι' αυτό, γιατί καταστρέφεται η χώρα τους είναι ένας δόκιμος πλέον όρος. Άρα, αφισχύει και για τους πρόσφυγες γενικότερα. Δηλαδή, να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες για να έρθουν στην Ευρώπη και να ζήσουν ελεύθερα μέσα σε κατάσταση απόλυτης ελευθερίας. Number 691. 691. Καλημέρα. Γέννης από τη Γερμανία. Δύο ερωτήσεις. Ζούμε στην Ευρώπη, ένα από τα πλουσιότερα μέρη της γης και βλέπουμε όμως τους στόχους μας για την προστασία του κλίματος να κατεβαίνουν όλο και περισσότερο. Κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ, όλοι σας οδηγείτε μεγάλα δυνατά αυτοκίνητα με πολλές εκπομπές διοξιδίων του άνθρακος. Γιατί προωθείτε τόσο λίγο την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων. Βρισκόμαστε εδώ στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, με πυρηνικά εργοστάσια και μάλιστα των οποίων η κατάσταση είναι τόσο επικίνδυνη που ομοσπονδιακά γερμανικά κρατήδια προσφέρουν στο δικαστήριο για να διακόψουν την ε, λειτουργία τους αυτά μονάχα για να αυξάνουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων που παράγουν ενέργεια και που καταστρέφουν, μπορεί ενδέχεται να καταστρέψουν κάποτε την ίδια την Ευρώπη. Ούτε 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος δεν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολύ κάτω από το μέσο όρο ολόκληρου του κόσμου. Εγώ το θεωρώ αυτό πραγματικά ένδειξη φτώχειας. Θα ήθελα να μάθω, αφού βρισκόμαστε εδώ, μια Ευρώπη έχουμε, ένα πλανήτη έχουμε. Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε τι ευκαιρίε που μα δίνουν οι στι πηγές ενέργεια. Ευχαριστώ. Και τελευταίο, απολύτω τελευταία ερώτηση, το 223. Ε, ονομάζομαι ε, Ρέι, είμαι φοιτήτρια και ασχολούμαι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στις ε, Βρυξέλλες. Μιλήσαμε για τον πρόεδρο Τραμπ και για τη Συμφωνία των Παρισίων. Επειδή η Ένωση βρίσκεται στο προσκήνιο των διαπραγματεύσεων, πώς θα προσπαθήσει να κρατήσει τις ΙΠΑ επίσης στο προσκήνιο μέσα στα πλαίσια ε, των ε, ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών. Πώς θα τους πιέσουμε ε, να συμμετάσχουν ενεργά στην Συμφωνία των Παρισίων, γιατί αν αποχωρήσουν μηδενίζονται όλα. Τώρα επανερχόμαστε τη σοφία των συναδέλφων. Ο κύριος Eichhout έχει πρώτος το λόγο. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να μιλήσω μόνο για δύο λεπτά γιατί τελειώ ε, θα με μαλώσει, θα χτυπήσει το σφυράκι. Όσον αφορά τι εμπορικέ συμφωνίε, ε, είναι σαφέ νομίζω ότι εγώ καταψήφισα την εμπορική συμφωνία με τον Καναδά και είναι σημαντικό να ρωτήσετε του ευρωβουλευτέ σα τι ψήφισαν. Βέβαια, ο αγώνα δεν έχει τελειώσει. Τώρα το θέμα θα πάει στα εθνικά κοινοβούλια και όλα θα αποφασίσουν τι θα γίνει με την εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Αυτή την ερώτηση είναι σημαντική να την κάνετε, να ρωτήσετε όλου του βουλευτέ βουλευτέ σα, γιατί εκκρεμεί ακόμα η ψηφοφορία. Αλλά είναι σημαντικό να μην πέσετε στην παγίδα να λέτε ότι το εμπόριο αυτό καθεαυτό είναι κακό. Δεν είναι έτσι. Είναι καλό. Αλλά ο τρόπο ε, με τον αντιμετωπίζουμε τώρα είναι κακό. Ε, δεν είναι καλή αυτή η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Υπάρχουν άλλε καλέ εναλλακτικές λύσει. Προ τον Ρικάρδο στην Πορτογαλία. Έχει απόλυτα δίκιο. Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Τι θα γίνει με τα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καμία χώρα εκτός από τη Σουηδία δεν καλύπτει τις διεθνείς της υποχρώσεις ε, να καταβάλει χρήματα ως ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Όλοι μιλάνε για τον Τραμπ και για τον ΝΑΤΟ και ξεχνάνε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις από το να μην πληρώνουμε για αναπτυξιακή βοήθεια. Στον Γέντσα από τη Γερμανία. Εγώ ποδήλατο χρησιμοποιώ. Τι να σα κάνω, δίκιο έχετε για του άλλου, αλλά εγώ ποδήλατο χρησιμοποιώ και να σα πω και κάτι. Επικίνδυνο το ποδήλατο στι Βρυξέλλε. Για τα πυρηνικά πρέπει να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιτρέπει ενισχύσει από την, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία για να κατασκευαστούν νέα πυρηνικά εργοστάσια. Τρελό αυτό. Νέε ενισχύσει για νέα πυρηνικά εργοστάσια και η Ουγγαρία μα καθιστά ακόμα πιο ε, εξαρτώμενους από τον Πούτιν. Και αυτό πρέπει να φυγεί. Τέλος, για τον Τραμπ Ράιντι νομίζω η Ινδία, η χώρα η οποία πέρασε στην πράσινη οικονομία, θα ε, προηγηθεί, θα χαράξει τον δρόμο και έτσι ε, θα μπορέσει να πείσει τον Τραμπ. Ε, αυτός μπορεί να κρατήσει τα παλιά ανθρακοριχεία, αλλά θα του δείξει το δρόμο και αργότερα ο Τραμπ και αυτός ε, θα αλλάξει γνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Λάινερ, Γιώ Κοιτάξτε, θα αλλάξει η εμπορική πολιτική. Θα αλλάξει η εμπορική πολιτική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. ΣΕΤΑ και ΤΙΤΙΠ είναι τα καλύτερα παραδείγματα. Και στο κοινοβούλιο στο μέλλον θα υπάρχει σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες μία ρήτρα βιωσιμότητας. Δηλαδή ε, θα εξετάζουμε τα περιβαλλοντικά, τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τα κοινωνικά κριτήρια και ε, Υπάρχει και καλό εμπόριο, ας πούμε, με ηλιακούς ε, συλλέκτες. Να μην υπάρχουν ε, φραγμοί. Η βιωσιμότητα θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Ε, το κλίμα θα είναι μεγάλο πρόβλημα, ήδη είναι σήμερα και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στους ετούντες άσυλο αυτό που δεν έκανε η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία δέχτηκε κάποιους από αυτούς, αλλά όχι η Αυστραλία. Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρική ε, κινητικότητα. Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στην τεχνολογία diesel, ε, από κάποιο πρίσμα καλή, από άλλο πάλι κακή για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Οι Κινέζοι προάγουν την, ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έχει έρθει η στιγμή πλέον και εμείς ε, να εστιάσουμε σε αυτό. Να έχουμε πράγματι μόνο 20% εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ε, εγώ έχω τη Γερμανία με τη Δανία, ίσως και τη Σουηδία. Είμαστε σκαπανείς σε αυτό το θέμα. Και Θέλω να πιστεύω ότι και άλλοι θα μας ακολουθήσουν, γιατί μετά από κάποια χρόνια θα είναι δωρεάν οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Για τη συντήρησή τους θα υπάρχουν δαπάνες, αλλά όχι για την ίδια την ενέργεια. Επιβιώσαμε με τον Μπούς, θα επιβιώσουμε και τον, με τον Τραμπ να είμαστε αισιόδοξοι. Um, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, καταρχήν γιατί παρευρεθήκατε εδώ στη συζήτηση. Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της Ευρώπης είναι να ακούμε ο ένας τον άλλον. Ήταν μακρύ το απόγευμα, αλλά ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον, αλλά και περίπλοκο γιατί υπάρχουν ε, πολλές απόψεις στις κλιματικές αλλαγές, ανεργία των νέων και ούτω καθεξής. Εμείς καθόμαστε στις δικές σας θέσεις και δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά θα πρέπει να βρούμε κοινό έδαφος και γι' αυτό μιλάμε για συμβιβασμούς. Η λέξη αυτή θεωρείται αδυναμία πολλές φορές στο σημερινό πολιτικό κόσμο. Όμως οι διαφορές θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμβιβασμούς. Πολλές φορές δεν γίνονται γρήγορα οι συμβιβασμοί και οι ερωτήσεις σας το αντικατοπτρίζουν αυτό. Σας ευχαριστώ όλους και τους συναδέλφους μου που συνεισέφεραν στη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πολλά μέλη δεν είχαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν. Έχουμε πολλά θέματα αυτή την εβδομάδα και τους ευχαριστώ που ήρθαν εδώ. Ευχαριστώ και το πάνελ που μας έδωσε νέες και καλές ιδέες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ταγιάννη που παρέμεινε στην αίθουσα αυτή. Ξέρω ότι έχετε πολλά θέματα που σας απασχολούν, αλλά ξέρω ότι αυτό το θέμα σας απασχολεί άμεσα μέσα στα πλαίσια της εντολής σας και σας ευχαριστώ που μείνατε εδώ μέχρι το τέλος της συζήτησης. Εγώ προέρχομαι από μία μικρή χώρα, την Ιρλανδία, και θα ήθελα να σας πω ότι και οι μικροί κάνουν τη διαφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουμε δει αυτό συνεργαζόμενοι και όταν γνωρίζουμε οι μεν τους δε τα καταφέρουμε όπως και στο σχολείο ή στον αθλητισμό. Πρόκειται για ένα μεγάλο χώρο, μεγάλο αριθμό, διαφορετικές γλώσσες, αλλά όλοι θέλουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Όχι μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά και για τις επερχόμενες γενές. Αλλά θα πρέπει να μας βοηθήσετε στην οικοδόμηση της Ευρώπης αυτής.